το μεσημέρι στις 12. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αύριο, Τρίτη, 15 Απριλίου, θα ξεκινήσουμε στις 8.30 το πρωί και θα συζητήσουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μετά θα έχουμε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε από τις 3 έως τις 11 το βράδυ. Την εμείς διάταξη μπορείτε να τη βρείτε στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κλείνει εδώ η σημερινή συνεδρία. Σας ευχαριστώ.